δεν θα πρέπει να συζητάμε αντισημιτισμό, ρατσισμό και απεριζόμαστε μόνο σε αυτό. Υπάρχει και η ανάγκη να δούμε ότι αυξάνεται ο αντισημιτισμός στην Ευρώπη και στην πατρίδα μου, στη Σουηδία. Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, ο αντισημιτισμό αυξάνεται σαν φαινόμενο κυρίως στη Σουηδία. Οι Εβραίοι δεν αισθάνονται πλέον ελεύθεροι να φοράνε το άστο του Δαβίδ ή το κύπα στο κεφάλι. Ε, πιστεύω ότι το έργο κατά του αντισημιτισμού θα πρέπει να έχει πολύ σαφέστερη προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν κατανοώ, διότι δεν αναφέρεται καν αυτή η πτυχή στο πρόγραμμα εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήθελα μία εξήγηση, μία απάντηση γιατί δεν υπάρχει αυτή η μνήα. Κλείνοντας, θα ήθελα να κάνω συγκεκριμένες προτάσεις πρωτοβουλία για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρώτη πρόταση, να αυξηθεί η χρηματοδότηση για την κατάρτιση, την εκπαίδευση των νέων όσον αφορά τη ΣΟΑ και τα εγκλήματα μίσου στην Ευρώπη. Δεύτερον, πρέπει να εγγυηθούμε το μπλοκάρισμα της χρηματοδότησης, εξωτερικής χρηματοδότησης του φονταμενταλισμού στην ε, Ευρώπη Τρίτον, πρέπει να εμποδίσουμε εκείνου που διαδίδουν το μίσο να μπορούν να έρχονται και να τριγυρνάνε στην Ευρώπη και να διασπείρουν αυτέ τι ακρεφνεί θέσει. Θα πρέπει να τεθεί τέρμα στον αντισημιτισμό και στο ρατσισμό στην Ευρώπη, διότι δεν θα πρέπει να ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο αυτά τα φαινόμενα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τα τελευταία χρόνια είδαμε ανησυχητικά σημεία περιπτώσει αντισημιτισμού στην Ευρώπη και στον κόσμο και στην πατρίδα μου στην Ιταλία πρόσφατα εμφανίστηκαν σύμβολα αντισημιτικά και διάφορες επιγραφές αναφερόταν στη ΣΟΑ και στράφηκαν κατά των ακτιβιστών κατά του φαινομόνου καλύπτεται από κόμματα που χρησιμοποιούν το ρατσισμό για να κερδίσουν ε, συνένεση. Οι ηγέτες αυτών δυνάμεων πολύ συχνά κάνουν δηλώσεις αντισημιτικές, καμιά φορά αρνούνται το ίδιο το ολοκαύτωμα. Εδώ και κάποιε εβδομάδε αυτό το κοινοβούλιο φιλοξένησε τη Γιάννα Σέγκρε που επέζησε του Auschwitz. Σήμερα χρειάζεται να ακολουθήσουμε το παράδειγμά τη, διότι αρνήθηκε την πρόσκληση για μη συζήτηση για τον αντισημιτισμό μαζί με εκπροσώπους της ακραία δεξιάς. Θα πρέπει να πούμε σαφώς ότι μόνο αν, είμαστε, αν είναι κάποιοι καθαρά αντιρατσιστέ μπορούν να καταπολεμήσουμε τον αντισημιτισμό. Σαν κοινοβούλιο θα πρέπει να είμαστε στην πρώτη γραμμή, να καταπολεμούμε όλα αυτά τα φαινόμενα. Και η αποκατάσταση ομάδα εργασία για τον αντισημιτισμό είναι ένα σημαντικό μήνυμα, αλλά θα πρέπει να δώσουμε συνέχεια προ αυτή την κατεύθυνση. Σα ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε. Κύριε Χακαράινεν τώρα. Μάλλον ο κύριο Χακαράινεν έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για να μην λησμονούμε την αλήθεια, πρέπει να πούμε ότι σύμφωνα με μια δημοσκόπηση λένε οι Εβραίοι ότι η βία και οι απειλές βιοπραγίες κατά αυτών διαπράτεται περισσότερο από τους μουσουλμάνους, κατά κύριο λόγο. Οι ακροδεξιοί και, και εκπρόσωποι της άκρας αριστεράς και αυτοί απειλούν τους Εβραίους. Βεβαίως πρέπει να κάνουμε κάτι για τον αντισημιτισμό αλλά σήμερα πάρα πολύ εύκολα κατηγορούνται κάποιοι ως ρατσιστές. Αν είναι κανείς εθνικιστής, πολύ συχνά λέγεται ότι είμαστε και ρατσιστές ως εθνικιστές. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία, μπορεί πάντα κανείς αβάσιμα να καλέσει κάποιον ρατσιστή. Και μπορούν να υπάρχουν λάθος ισχυρισμοί. όσον αφορά τι κατηγορίε ότι είναι κάποιο ρατσιστή. Είναι πολύ εύκολο να επιτίθεται κανεί κατά ανθρώπων και να του αποκαλεί εθνικιστέ. Και καμιά φορά τα δικαστήρια παίζουν το παιχνίδι αυτό και τα δικαστήρια τιμωρούν κάποιου που θεωρούνται ω ρατσιστέ παρά μόνο που είναι μόνο εθνικιστέ. 75 χρόνια πέρασαν από την απελευθέρωση του Auschwitz και όλοι είπαμε ότι δεν πρέπει να ξανασυμβεί ποτέ αυτό. Δυστυχώ, όμως υπάρχουν επαναλήψεις και στα Βαλκάνια και με τους Τούτσι, με τους Κούρδους, τους Κόπτες, τους Φαλασσά, τους ε, Ινδούς, Μουσουλμάνους, τους Παλαιπιστινίους, τους Ρώμα κλπ. κλπ. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε ξανά τον αγώνα μας και πώς θα αντιμετωπίσουμε τα φαινόμενα αυτά σωματικά και ψυχικά. Η κατάσταση δεν ε, συγκρίνεται. Πρέπει να υπάρχει ε, η ειδική ρητορική η οποία να μην διχάζει αλλά να ενώνει. Η πρόκληση είναι μεγάλη. Χρειάζεται αλληλεγγύη και προσπάθεια από όλου για όλου. Πρέπει να δεσμευτούμε κατά των διακρίσεων οικουμενικά, χωρί να σκεφτόμαστε την προέλευση, το φύλλο, τον ε, σεξουαλικό προσανατολισμό ή οποιοδήποτε άλλο κριτήριο που μπορεί να χαρακτηρίζει κάποιον. Δεν χρειάζεται να είναι κανεί γυναίκα για να υποστηρίζει τη γυναίκα, ούτε να είναι ε, Εβραίο, Χριστιανό ή Μουσουλμάνο για να στηρίξει έναν Εβραίο, Χριστιανό ή Μουσουλμάνο, ή ομοφυλόφιλο για να στηρίξει έναν ομοφυλόφιλο. Είμαστε όλοι ανθρώπινα όντα και δεν χρειαζόμαστε διακρίσει. Ευχαριστούμε. Βόιντρα Αλεξάνδρα τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Πιστεύω ότι όταν κοιτάμε τα ε, νούμερα και τι έχει γίνει με τον αντισημιτισμό, ε, βλέπουμε πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα. Πριν από 10 χρόνια, 60.000 έφυγαν από τη Γαλλία και η Υπηρεσία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων λέει ότι 30% των ε, Εβραίων σκέφτεται να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά τα νούμερα είναι φοβερά. Στη Γερμανία επίσης είναι κοντά στο 40%, 30% στη Σουηδία και αυξάνεται τα τελευταία χρόνια. Ε, Γαλλία 44%, Βέλγιο όπου και εκεί Επίση, ε, περνάμε πολύ χρόνο τη ζωή μα. Μεγάλο το Ουγγαρία. Η Ουγγαρία είναι η μόνη χώρα η οποία έχει μειώσει τον αριθμό των Εβραίων που φεύγουν από τη χώρα. Είναι περίπου στο 10%. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν, να ε, δούμε καλύτερα τον ορισμό του αντισημιτισμού, να πολεμήσουμε τη Χεσμολά και να σταματήσουμε επιτέλους με αυτές τις εξωτερικές πολιτικές που μας ζημιώνουν τόσο. Η κυρία... Αγαπητέ συνάδελφε, δέχεστε μία γαλάζια κάρτα. Δέχεστε μπλε κάρτα, αγαπητέ συνάδελφε. Δέχεστε την μπλε κάρτα. Ναι. Ο κύριος Πόλτσακ. Ευχαριστώ. Αγαπητέ συνάδελφοι που δεχτήκατε την μπλε κάρτα. Άκουγα την ομιλία και πήρετε από το στόμα μου αυτά που θέλω να πω. Αλλά θέλω να πω ότι ο ρατσισμός δεν είναι απλά αντισημιτισμός. Γιατί εσείς αναφερθήκατε μόνο στον αντισημιτισμό, δηλαδή ρατσισμό σε βάρος των Εβραίων, αλλά υπάρχουν και άλλες μορφές ρατσισμού. Τις θεωρείτε και αυτές πολύ σημαντικές μορφές ρατσισμού. Απάντηση. Ναι, βεβαίως. Απλά ο αντισημιτισμός λόγω της ιστορίας ε, της Υπήρου, το τι γινόταν ε, τον 20ο αιώνα, κατά την άποψή μου είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Και αν δει κανεί και τα νούμερα, είναι σαφές ότι είναι τεράστιο το πρόβλημα. Και σχετίζεται με τη μεταναστευτική πολιτική, κάτι που δεν πρέπει να αποκρύπτουμε, και την πολιτική ρητορία. Αν δείτε τα στοιχεία, θα δείτε ότι έχουμε αυτούς τους 60.000 ανθρώπους που δεν νιώθουν άνετα και θέλουν να φύγουν. Ευχαριστώ. Κυρία Σημακοπούλη. Κύριε Πρόεδρε, την τελευταία δεκαετία ο αντισημιτισμός αύξησε, σήκωσε το άσχημο κεφάλι του στην Ευρώπη. Δυστυχώς αυτό στηρίζεται και με στοιχεία. Σύμφωνα με το Ρωμανόμετρο το 2019 υπάρχει τεράστια διαφορά στον αφορά την αντίληψη του αντισημιτισμού. Περίπου 90% των Εβραίων αισθάνονται ότι αντισημιτισμό αυξάνεται, αλλά μόνο 36% των Ευρωπαίων πολιτών συμφωνούν. Η Ευρώπη δεν μπορεί να επιτρέψει το δηλητήριο του αντισημιτισμού να διαδοθεί. Πρέπει να προστατεύσει, να υποστηρίξει τους Εβραίους της και θα πρέπει αποτελεσματικά να καταπολεμήσει εκείνους που διαπράττουν δυσημιτικές πράξεις. Και αναμφισβήτητα το Χεσμολά που είναι εκπρόσωπος του, θανατηφόρος του Ιράν είναι η πιο ε, σοβαρή απειλή κατά των Εβραίων στην Ευρώπη και όχι μόνο στην Ευρώπη. Όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση αρνείται ε, να ακολουθήσει τα βήματα κάποιων από των πλών αγαπητών συμμάχων όπως είναι η ΕΠΑ, όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, όπως είναι ο Καναδάς, και να θέσει τέρμα σε αυτή την ψευδή διάκριση μεταξύ πολιτική πτέρυγα και στρατιωτική πτέρυγα του Χεσμολά. Μια διάκριση που ηρίστον παρόδο αποκαλεί αστείο και απορρίπτει ο Χεσμολά. Αυτή η υποκρισία θα πρέπει να σταματήσει τώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να βάλει το Χεσμολά στο σύνολό του στην λίστα τρομοκρατικών ομάδων της Ευρωπαϊκής Ενώσης αν θέλει να είναι αξιόπιστη και πιο σημαντικό αποτελεσματική στην καταπολέμηση του αντισημιτισμού και των φρικαλαίων πράξεων που είναι αποτέλεσμα του αντισημιτισμού. Σας ευχαριστώ. Κυρία Σίλβια Σπούρεκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως ήδη ακούσαμε, το διάφορες έρευνες και το γυροβαρόμετρο δείχνουν ότι η συμμετική ε, βιοπραγία αυξάνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύντομα με την, με την έρευνα του ΦΡΑ δεν μπορούν να ζήσουν ελεύθεροι χωρίς ανησυχία οι άνθρωποι. Ανησυχούν για την ασφάλεια τη δική τους και των μελών της οικογένειάς τους. Αλλά ο ρατσισμός και ο αντισημιτισμό εξακολουθούν να απορρίπτονται από διάφορους πολιτικούς μέσα ενημέρωσης και επιστήμονες σε όλη την Ευρώπη. Όταν ήμουν υπεύθυνοι για ανθρώπινα δικαιώματα, ε, σαν επίτροπος άκουγα να λέγεται ότι δεν υπάρχει αντισημιτισμός στην Πολωνία, ενώ αντιμετώπιζα λόγους μισολοδοξίας και βιοπραγίες κατά των Εβραίων. Είναι 21ος αιώνα και όλο και περισσότεροι εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση αισθάνονται ότι μπορούν να αντιμετωπίζουν κάποια διαφορετικά και να τον μισούν τον άλλον λόγω της θρησκείας του, της ή τη προέλευση του τη ή του χρώματο τη επιδερμίδα του τη. Είναι απαράδεκτο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατεπηγόντω χρειάζεται μια στρατηγική κατεπολέμηση του του ρατσισμού, τη ξενοφοβία για να προλάβει και να καταπολεμήσει αυτά τα φαινόμενα, να προστατεύσει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σα ευχαριστώ. Our next... Δέχεστε την γαλάζια κάρτα, κυρία Ορίστε. E, e, Έχω μια ερώτηση απευθυνόμενος προς συνάδελφο. Όταν ήσασταν υπεύθυνοι σαν συνήγορος του πολίτη θυμόσαστε πώς αντιδρούσε η αστυνομία όσον αφορά τα διάφορα αντισημετικά ε, επεισόδια. Ήμουν υπουργό Εσωτερικών στην κυβέρνηση νόμου και δικαιοσύνης και οποιοδήποτε σημάδι αντισημιτισμού καταπολεμεί το από την αστυνομία. Δεν υπήρξε παραδοχή, πάντα υπήρχε αντίδραση για τον συμμετισμό. Μην παραπλανείτε λοιπόν το κοινοβούλιο με αυτά που λέτε. Δύο λάθη κάναμε. Επειδή είχατε μιλήσει κανονικά δεν έπρεπε να είχατε ζητήσει ε, την ε, μπλε κάρτα και το δεύτερο λάθος ήταν ότι δεν κάνατε καν ερώτηση, ε, τέλος πάντων. Παρ' όλα αυτά, ε, η κυρία Σπούρεκ νομίζω θέλει να απαντήσει, οπότε της δίνω τη δυνατότητα αυτή. Ναι, ευχαριστώ. Θέλω να απαντήσω. Τη μία ερώτηση. Και να πω ότι δεν αρκεί να τη δράσει νομία. ή εισαγγελεί να διώκουν και τα δικαστήρια να δικάζουν. Δεν είδα το βαθμό της αποφασιστικότητας που θα ήθελα τουλάχιστον να. Ήμουν αναπληρώτρια συνήγορος του πολίτη στην Πολωνία και πρέπει να σας πω ότι χρειάζεται η καταγγελία από τα υψηλότερα κερμάκια της κυβέρνησης. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γκαγό έχει τώρα το λόγο. Το θέμα που συζητάμε σήμερα συζητιέται συχνά εδώ στο Μικύκλιο και καλά κάνει. Αλλά το αντιμετωπίζουμε με ελλειπή τρόπο και με μονόδρομο. Γιατί εδώ κανείς, η πλειοψηφία τουλάχιστον, δεν ασχολείται με τις δράσεις κατά των χριστιανών ανά τον κόσμο, όπου πλήττονται περιουσίες αλλά και εκκλησίες. Οι περισσότεροι εδώ πέρα ευρωβουλευτές δεν θέλουν να θέσουν το πραγματικό ερώτημα αυτό που ενοχλεί, που πειράζει. Ποιος είναι ο κύριος λόγος, η κύρια αιτία της αύξησης των δράσεων αυτών κατά των Εβραίων και κατά των Χριστιανών. Μα την ξέρετε την απάντηση, είναι η άνοδο του Ισλαμισμού, του ολοκληρωτισμού αυτού που αρνείστε να δείτε, που δεν επικρίνεται ενώ τον υφίστανται οι λέει μα. Όσον αφορά το μίσο, εδώ κάνετε λάθο. τα βάζετε πάντα με αυτούς που ονομάζετε λαϊκιστές. Όχι, τις προσπάθειές σας πρέπει να τις στρέψετε σε αυτούς που μισούν τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, τις ατομικές μας ελευθερίες. Πρέπει να αγωνιστείτε κατά αυτών που θέλουν βία να μας επιβάλλουν μια βάρβαρη κοινωνία που δεν είναι η δικιά μας. Αυτός πρέπει να είναι ο κοινό μας αγώνας. Με όλες μας τις δυνάμεις να καταπολεμήσουμε τον Ισλαμισμό, τον ριζοσπαστικοσμό, το, που είναι η μεγαλύτερη απειλή που βαραίνει πάνω στις δημοκρατίες του 21ου αιώνα. Ευχαριστώ. Χέλμουτ Κόικινγκ. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Πραγματικά με αυτά που ακούω εκπλήσωμαι. Φαίνεται ε, ότι είναι ε, το πιο αποτρόπαιο πράγμα που έχει γίνει στη, στον κόσμο ο αντισημιτισμός ε, και έχουμε αυτή τη νέα τάξη στη δημοκρατία ε, που έχει, ε, έχουν, έχει χάσει πολλά, αλλά ο αντισημιτισμός όχι, ισχύει ακόμη. Και φαίνεται ότι είναι κάτι ριζωμένο βαθιά στην κοινωνία. Το δείχνει και η κοινωνία. Έχουμε τις λαϊκιστές της δεξιάς. Ε, πολλές φορές δεν κάνουν καν διακρίσεις και πολλές φορές... Ε, ε, φυτεύουν τον αντισημιτισμό ε, στο μυαλό των ανθρώπων ε, με αυτά τα οποία λένε και υπάρχει κοινικό, κοινική περιφρόνηση. Όλο αυτό θα πρέπει να το εκριζώσουμε από τον πολιτικό τοπίο και από την κοινωνία και θα πρέπει και τον αντισημιτισμό να τον ακριζώσουμε. Χρειάζεται μια νέα νοοτροπία γιατί δεν έχουμε ανάγκη από άλλους ήρωες ε, στις χώρες. Ε, όλοι πρέπει να καταδικάσουμε αυτά τα φαινόμενα. Ευχαριστώ, Εμίλιο Νούνο. Ευχαριστώ. Η συζήτηση αυτή κατά του αντισημιτισμού θυμάμαι τι έγινε στο Πορντό όπου ένας Πορτογάλος έσωσε ένα σωρό Εβραίους οι οποίοι ξέφευγαν από τον ναζισμό. Είμαστε μια ουδέτερη χώρα, υπήρχαν οι οδηγίες από την κυβέρνηση, σταμάτησαν να δίνουν θεωρήσεις στους Εβραίους. Προσπαθήσαμε να μην κάνουμε διακρίσεις. Το τίμημα που πληρώσαμε βέβαια ήταν πολύ μεγάλο διότι απαγορεύτηκε στον άνθρωπο αυτό να σκίσει πλέον τα... τη δουλειά του, το επαγγελμά του. Κατέληξε στη φτώχεια. Και κυκλοφορούσε με ρούχα ελεημοσύνης που του δίνανε δεξιά και αριστερά. Ε, τελικά ε, τιμήθηκε βέβαια αργότερα και αναφέρθηκε αυτή η συνεργασία. Στην Πορτογαλία, μετά το θάνατό του βέβαια, ε, του αποδόθηκαν διακρίσεις. Αξίζει σε παγκόσμιο επίπεδο αναγνώριση ο άνθρωπος αυτός. Έδειξε ανθρωπισμό και μας εμπνέει εμάς και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και εγώ που είμαι Δημοκράτης και Πορτογάλος ήθελα να του αποδώσω φόρο τιμής εδώ. Κόλας, ε, Λούκας Κόχουτς Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Πριν από 75 χρόνια μετά το ολοκαύτωμα, ο αντισημιτισμός, το μίσος, οι διακρίσεις, η ξενοφοβία εξακολουθούν να αυξάνονται στην Ευρώπη και στην δικιά μου τη χώρα, στην Πολωνία. Ε, υποφέρουν και καταδίκα στο κοινοβούλιο την κοινότητα των ΛΟΕΤ. Εγώ δεν ανήκω σε αυτή την κοινότητα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορώ να μείνω αδιάφορος διότι η αδιαφορία είναι αυτή που πειράζει, που πλήττει τη δημοκρατία, την ελευθερία και την ελεγγύη. Επίσης πιστεύω, αν ήμουν εγώ στη θέση τους, τι θα γινόταν. Ε, Μάριον Τούλσκι, ε, που επέζησε από το ολοκαύτωμα είπε ακριβώ ότι η ΣΟΑ δεν έπεσε από τον ουρανό, αλλά δημιουργήθηκε βήμα-βήμα, σιγά-σιγά και βασίστηκε στις διακρίσεις και κατέληξε στα στρατόπεδα ε, συγκέντρωσης και αφανισμού. Ο κόσμος αυτά πρέπει να τα θυμάται και να μην επαναληφθούν ποτέ. Και ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να αγωνιστούμε κατά οποιαδήποτε μορφής μίσους και διακρίσεως. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκολας Φέστ. Ευχαριστώ πολύ. Το βασικό μας πρόβλημα είναι ότι ε, ακούμε πράγματα ανέσχυντα. Μιλάμε για η κυρία Ρίσπαρντος χάρη, μιλάει ε, για ε, Εβραίους που ε, θανατώνονται αλλά δεν λέει το όνομα ε, του θήτη ή δεν λέει ότι ήταν ένας μουσουλμάνος ε, που είχε μεταναστεύσει και αναφέρουμε άλλες τρομοκρατικές οργανώσεις, δεν αναφέρουμε τη Ε, και όταν ανοίξαμε τα σύνορα με, τη την και το Παγκόσμιο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση, ανοίξαμε τα σύνορα σε περισσότερους ε, μετανάστες ε, ε, και λένε οι Εβραίοι, παραδείγματος χάρη στο Βερολίνο, ότι οι περισσότερες επιθέσεις προέρχονται από μουσουλμάνους. Παρ' όλα αυτά, μουσουλμάνοι χρηματοδοτούνται. Οι Φατάχοι Χαμάς χρηματοδοτούνται με 1,5 εκατομμύρια την μέρα, είπε ο κύριος Μπορέλα. Αν λοιπόν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τον αντισημιτισμό, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να σταματήσουμε τη χρηματοδότηση αυτή. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Πρόεδρος. Αυτό που είπατε για ανέσχυτα πράγματα, σας παρακαλώ να μην χρησιμοποιείτε αυτές τις ε, διατυπώσεις ε, εδώ σε αυτό το σώμα. Ε, και τώρα θα δώσω το λόγο στους υπόλοιπους συναδέλφους με πρώτη την κυρία Ντυπών. Αξιότιμε πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι, έχουμε την πρώτη συζήτηση σε αυτή τη θητεία για τον αντισημιτισμό στο Κοινοβούλιο. Ε, και υπό ε, τις ε, τραγικές επιπτώσεις ε, στο Χάλε. Πριν από δύο εβδομάδες ορτάσαμε την απελευθέρωση του Auschwitz και πραγματικά καταλαβαίνουμε με όλα αυτά ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε τον αντισημιτισμό. Πρέπει να δοθεί τέρμα. Ο αντισημιτισμός, ο ρατσισμός, εγκληματικά τα μίσους αυξάνουν. Δεν θα πρέπει να δώσουμε λιγότερη προσοχή. Δεν θα πρέπει να στρέψουμε αλλού το βλέμμα. Και ακόμα πιο σημαντικό από το να στρέψουμε την προσοχή μας είναι να αντιμετωπίσουμε αυτό το διχασμό και την ε, ρητορική μίσους. Ε, έχουμε δει πάρα πολλά ε, πράγματα που δεν αντιμετωπίζονται ως αξιόπινες πράξεις, ενώ είναι και αυτό δεν αλλάζει, δεν βελτιώνει την κατάσταση. Θα πρέπει λοιπόν να πάρουμε πιο σοβαρή υπόψη την κατάσταση των θυμάτων, απειλέ, αντισημιτισμό στο διαδίκτυο και όχι να τον αντιμετωπίσουμε και να έχουμε ένα υψηλότερο επίπεδο φιλοδοξία. Μόνο ο ενωμένοι όλοι μαζί μπορούμε να σταθούμε απέναντι σε αυτό το φαινόμενο. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γιωκεβιτσιένε. Ο αντισημιτισμός είναι μια διάγνωση, μια σοβαρή ασθένεια τη κοινωνία. Όμως, για να βρει κανεί την σωστή θεραπεία, πρέπει να γνωρίζει τις αιτίε. Και ποιες είναι, είναι εσωτερικές και εξωτερικές αυτές οι αιτίες. Οι εσωτερικές είναι σαφείς. Είναι σαν μεταλλαγμένους ιούς, οι οποίοι ενεργοποιούνται σε ένα βρώμικο περιβάλλον ε, μίσους και εθνικισμού. Και αυτούς πρέπει να ξεριζώσουμε. Οι εξωτερικές αιτίε τώρα είναι οι διπλοπρόσωποι πολιτική του Κρεμλίνου σε βάρος της Ευρώπης. Και από τη μία τα βάζουμε τις χώρες ε, που λένε ότι είναι αντισημιτικές και ε, θέλουν, λένε, να καταπολεμήσουν τον ναζισμό. Από την άλλη μεριά όμως χρηματοδοτούν εθνικιστικά κόμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόταση του Πούτιν για να υπάρξει θέση ε, μόνιμη στο Συμβούλιο Ασφαλείας κατά του αντισημιτισμού είναι μια κοροϊδία γιατί η Ρωσία η ίδια αναβιώνει τον ολοκληρωτισμό του Στάλιν. Ο αγώνας κατά του αντισημιτισμού πρέπει να είναι κάτι στα πλαίσια της αποκατάστασης των ε, καθεστώτων του ολοκληρωτισμού σύμφωνα με τους Ρώσους. Αγαπητοί συνάδελφοι, γίνεται αυτή η συζήτηση διότι παρατηρούμε μια αύξηση του αντισημιτισμού και του ρατσισμού ε, και του μίσου στην Ευρώπη και παρακίνηση σε πράξεις ε, μίσου. Δεν θέλουμε περαιτέρω κλιμάκωση. Ξέρουμε ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε πολιτική εκμετάλλευση, όπως έγινε κατά το παρελθόν από τους δικτάτορες. Το 81% του εβραϊκού πληθυσμού σήμερα στην Ευρώπη ε, εκφράζει ανησυχίε όσον αφορά τον αντισημιτισμό. Και αυτό αφορά και την κεντρική και ανατολική Ευρώπη, όπου ο μουσουλμανικός πληθυσμός είναι πάρα πολύ μικρό σε ποσοστό. Στην Πολωνία, πράγματι, η αντίληψη για τον αντισημιτισμό είναι κάτι που δέχονται 48% του πληθυσμού, 42% στην Ουγγαρία. Για να αντιταχθούμε σε αυτές τις ρατσιστικές ε, παρενέσεις ε, και το μίσος έναντι των ανθρώπων, εναντίον της ανθρώπινης αξιοπρεπίας, είναι απαραίτητο να ξέρουμε την ιστορία για να το πετύχουμε αυτό και να εκπαιδεύσουμε τους ανθρώπους και χρειάζεται μια διοντολογική παιδεία ε, καταπολέμηση της μυσαλλοδοξίας. Αυτές ε, οι ομιλίες μίσους δεν πρέπει να γίνονται ανεκτέ, όπως έλεγε και αντιπρόεδρος τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παράδειγμα που θα μπορούσε να είναι παράδειγμα συγκεκριμένο αφορά μια ομιλία ε, μίσου του Καρδιναλίου Ντούκα κατά του μίσους που εξεφράστησε που είχε εκφράσει κάτι ε, που δεν ήταν τόσο καλό όσον αφορά τους ε, μουσουλμάνους. Κύριος Αντάμοβιτς έχει το λόγο. Ε, κυρία Ανταμοβιτ. αναφέρθηκαν πολλά. Αναφέρθηκε αυτό που είπε Μάριον Τούρσκι, που επεβίωσε του Auschwitz. Μας έδειξε από πού προήλθε το Auschwitz. Δεν έπεσε από τον ουρανό. αναφέρθηκε στα σημάδια ένας αποκλεισμός, αποξένωση, σταδιακός ε, και τελικά βιοπραγίες μέχρι το τελικό ε, βήμα της εξολόθρευσης. Δυστυχώς αυτό που μας είπε ε, είναι φρικτά επίκαιρο. Η σιωπηλή αποδοχή πάντα οδηγεί σε τραγωδία. Γι' αυτό όλοι είμαστε υπεύθυνοι. Όχι μόνο εκείνοι οι οποίοι το, σπέρνουν το μίσος, θα πρέπει και αυτοί να συνέλθουν, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε παθητικοί και να παρακολουθούμε τα τεκτενόμενα. Πρέπει να δράσουμε αποφασιστικά. Αν εξακολουθούμε να σιωπούμε, συμφωνούμε ότι αργότερα τα πράγματα θα έχουν προχωρήσει και θα είναι πολύ αργά. Ο Τούρσκι απίφθηνε έκκληση σε όλου ανεξαρτήτως θρησκεία ή θεώρηση θεώρησης των πραγμάτων. Δεν θα πρέπει να είσαι αδιάφορο, Ε, ου αδιαφορήσει είναι η ενδέκατη εντολή. Ε, λοιπόν, θα, θα πρέπει να κινούμεθα όταν παραβιάζονται δικαιώματα. Θα φανταστούμε έναν κόσμο που θα μπορεί να υπάρξει χωρίς μίσο. Σας ευχαριστώ πολύ. Τον επόμενο που θέλω να ευχαριστήσω για την πρωτοβουλία του ε, για την παρουσίαση μιας πρωτοβουλίας που κάνετε κατά τη Σιμψούν. Κύριε Βαντάλε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Πριν από 75 χρόνια είχαμε το Auschwitz Παρ' όλα αυτά παραμένει το μίσος στην Ευρώπη. Η οργάνωσή μας ε, καταγράφει διάφορα επεισόδια σε βάρος των Εβραίων και έχουμε καταλήξει ότι το 2019 1.800 τέτοια επεισόδια υπήρξαν στην Ολλανδία, που είναι το υψηλότερο, ο υψηλότερος αριθμός από ποτέ. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο μίσους κατά των Εβραίων. Η συναγωγή στην άλλη εδώ, στο Στρασβούργο πριν από τόσα χρόνια, είχε επίση μια επίθεση. Και συνεχίζονται αυτές οι δράσεις μίσους. Και ακόμα και στο εργατικό κίνημα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και η κυρία Μιρέγι Κνόλ στη Γαλλία δολοφονήθηκε στο διαμέρισμά της στο Παρίσι. Αλλά και στη δικιά μου τη χώρα έχουμε διάφορα τέτοια επεισόδια. Φτάνει πια ο αντισημιτισμός. Στηρίξτε το www.stopantisemitism.eu. Πρόκειται για μια συλλογή υπογραφών. Υποστηρίξτε μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Μπάλας Χιτβέγγι είναι επόμενος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σημαντικό θέμα και πρέπει να διατυμπανίσουμε ότι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η μόνη αντιμετώπιση στον αντισημιτισμό είναι η μηδενική ανοχή. Στην Ουγγαρία η κοινωνία, οι πολιτικοί συμφωνούν απόλυτα. Τα μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ζουν σε ασφαλείς συνθήκες, μπορούν να ασκούν τη λατρεία τους, να ζουν ελεύθερα, γιατί το σύνταγμά μας, αλλά η δική μας υποχρέωση επίσης, είναι η ανεξθρησκεία και η εβραϊκή κουλτούρα ανθεί, ε, αναβιώνει ε, στη χώρα μας. Ζουν ε, οι Εβραίοι ασφαλώς και κρατούν τις παραδόσεις τους. Ταυτόχρονα στη Δυτική Ευρώπη τα βία εγκλήματα σε βάρος μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας αυξάνονται. Πρέπει να σταθούμε απέναντι σε αυτό το φαινόμενο, αλλά και να συζητήσουμε ε, για να εξηγήσουμε το πώς ε, συνεισφέρει ε, αυτή η αντιμουσουλμανική επίσης ρατσιστική συμπεριφορά σε αύξηση των αντισημιτιστικών κρουσμάτων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κοκαλάρη. Έχει τώρα το λόγο. Πρέπει με σοβαρό τρόπο να αποθήσουμε τις διακρίσεις, το μίσος, το ρατσισμό. Προβλήματα στα οποία εκτίθενται οι Εβραίοι. Είναι εξαιρετικά ευάλωτοι οι Εβραίοι στη Σουηδία. Δέχονται επιθέσεις σε διάφορους τόπους από εξτεμιστές της, αρισ... δεξιάς, Ισλαμιστές και εκείνους που μισούν το κράτος του Ισραήλ. Οποιοςδήποτε ψώνει τη φωνή του Φοβάται. Δεν εκδηλώνουν τη θρησκεία του ανοιχτά. Φοβούνται διάκριση τα παιδιά των Εβραίων στο σχολείο. Ποιο δρά όταν ε, δέχονται επιθέσει ε, ε, οι συναγωγέ. Όχι η Σουηδική κυβέρνηση. Εγώ θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Ένωση να δράσει για να προστατεύσει του Εβραίου στην Ευρώπη. Θα πρέπει να εκπαιδεύουμε περισσότερο του νέου στα σχολεία και θα πρέπει να επενδύσουμε τόσο ώστε να υπάρχουν ευρωπαϊκοί νόμοι για να μποροκάρουν τη χρηματοδότηση εκείνων που είναι εξτρεμιστέ και που διαδίδουν αξίες αντιδημοκρατικές. Αρκετά μέχρι τώρα. Ευχαριστώ. Πηγαίνουμε στη δικασία Κατσιά, αλλά καταρχάς θα δώσω το λόγο στον κύριο Αντέμοφ. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Σήμερα καταγγέλουμε τις πράξεις αντισημιτισμού και ρασισμού λόγω εθνικότητας, εθνικής καταγωγής και θρησκευτικού μίσους. Κάτι βέβαια κατανοητό, διότι τέτοιες ενέργειες δεν έχουν κανένα χώρο εδώ. παρόλα αυτά θα πρέπει να κοιτάξουμε πολύ καλά στον καθρέφτη και να διερωτηθούμε κατά πόσον μπορούμε να ζητήσουμε τις τους ψηφοφόρους μας να υιοθετήσουμε μια πολιτισμένη στάση και προσέγγιση, αν όμως είμαστε και εμείς το καλό παράδειγμα ένας Έλληνα συναδελφός έσκησε τουρκική σημαία στο Μικύκλιο την προηγούμενη ε, Ολομέλεια. Εδώ, στο Λίγον τη Δημοκρατία, Είναι αυτό παράδειγμα σεβασμού και σωστή συμπεριφορά ή είναι πράξη μίσου. Εμεί, τα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου έχουμε το δικαίωμα να ε, φερόμαστε έτσι απέναντι σε ένα εθνικό σύμβολο μια χώρα, οποιασδήποτε, όχι τη Τουρκία συγκεκριμένα, οποιασδήποτε. Και γι' αυτό πριν ε, ζητήσουμε από ψηφοφόρου ή φίλου να μην είναι η συμπεριφορά του αντισημιστική, ρατσιστική κτλ., θα πρέπει εμεί να δώσουμε το παράδειγμα με μια πολιτισμένη ευρωπαϊκή συμπεριφορά. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε πολύ. Εδώ ολοκληρώθηκαν οι ε, παρεμβάσεις ε, και περνάμε στη σε Catch the Eye, όπως είπα και πριν. Ο κύριος Χέτμαν είναι ο πρώτος στον κατάλογο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε κυρίες και κύριοι. Πριν από λίγο καιρό γιορτάσαμε τότε την απελευθέρωση από το στρατόπεδο του Auschwitz. Τα τραγικά γεγονότα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου θα έπρεπε να είναι ένα καλό μάθημα για όλους και όλοι να τα θυμούνται. Δυστυχώς όμως κανείς δεν μπορεί να πει ότι τώρα στις αρχές του 2020 δεν υπάρχει στην υπηρό μας αυτή η ασθένεια του αντισημιτισμού, του ρατσισμού και του μίσους. Παρά τα γεγονότα που ζήσαμε πριν από λιγότερο από έναν αιώνα. Έχουμε την εσωτερική αγορά, έχουμε την ελεύθερη διακίνηση, αλλά να θυμόμαστε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργήθηκε κυρίως για να διατηρήσει την ειρήνη και να αποφύγει νέες συγκρούσεις και για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της υγείας, της δικαιοσύνης, της ελευθερίας. Είναι υποχρέωσή μας να προστατεύουμε αυτές τις αρχές. Οι κυβερνήσεις μας και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να φροντίζουν να ε, ξαφανίζουν κάθε δείγμα αντισημιτισμού, ρατσισμού και μίσους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο αντισημιτισμός, ο ρατσισμός και το μίσος στην Ευρώπη, λέει ο κύριο Μπλέξ, είναι πάρα πολύ βασικό και σοβαρό στοιχείο στην Ευρώπη. Εδώ όμω δεν περιγράφουμε μόνο την ιστορία, αναγνωρίζουμε σύγχρονες μορφές αυτών των φαινομένων. Σήμερα σκεφτόμαστε ότι μόνο κάποιοι ηγέτες ε, που προσπαθούν να χειραγωγήσουν την κοινή γνώμη είναι υπεύθυνοι. Τα στερότυπα προκαταλήψεις μπορούν να δημιουργήσουν ολόκληρη φωτιά, πυρκαγιά βάσει της ε, υπηκότητας. Για παράδειγμα στην Ιταλία ε, κάποιοι, υπάρχει μια περιοχή που ζουν ε, σλοβενική καταγωγή άνθρωποι, εκεί λοιπόν υπήρχαν διάφορα, ε, γράφανε στου τοίχου συνθήματα κατά αυτών. Ελπίζω η Ιταλική κυβέρνηση να το αντιμετωπίσει και να καταγγείλει αυτή τη συμπεριφορά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση από την πλευρά τη έχει μεγάλη ευθύνη για να αντιμετωπίσει κάθε τέτοια μορφή. Ευχαριστώ. Παίρνω το λόγο διότι οποιαδήποτε κίνηση αντισημιτισμού ή ρατσισμού ή μίσους, οποιαδήποτε εκδήλωση αυτών, δεν πραγματοποιούνται μόνο από μία μειονότητα. Είναι ένα κοινό πρόβλημα στην Ευρώπη. Πώς μπορούμε να λύσουμε αυτά τα προβλήματα. Να δώσω ένα παράδειγμα από τη χώρα μου, τη Βουλγαρία. Η ο Βαλέρη Σιμεώνοφ, ακραίο ακρεφνής εθνικιστής, εξελέγει σαν πρόεδρος του Κοινοβουλίου με την υποστήριξη του Βουλγαρικού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Αυτό είναι ένας άνθρωπος που προσπάθησε να στείλει πίσω ανθρώπους στα σύνορα με την Τουρκία που είχαν έρθει για να επισκεφθούν ή να ψηφίσουν ή να επισκεφθούν του συγγενείς τους. Κυρίε και κύριοι, δεν πρέπει να παραμένουμε σιωπηλοί, διότι το κακό μπορεί να έρθει και σε εμά μια μέρα. Θα πρέπει να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπειά μας. Θα πρέπει να διαφυλάξουμε τις ελευθερίες όλων των πολιτών. Με μικρόφωνο παρακαλούμε ο αντισημιτισμός, το μίσος ε, αξαπλώνονται στην Ευρώπη. Οι συζητήσεις ε, είτε στο δρόμο η καθημερινότητα είναι όλο και πιο επιθετικές ε, και προσβλητικές. Και στη Γερμανία βλέπουμε τις συζητήσεις πώς διεξάγονται. Αυτό πραγματικά είναι πρόσφορο έδαφος και για αντισημιστικές επιθέσεις που αυξάνονται σε βάρος ανθρώπων άλλου χρώματος, άλλης θρησκείας, μαύρους, Εβραίους, Ρωμά, Σίντι, που είναι στο στόχο της ρατσιστικής βίας. Στο Χάλε είχαμε την επίθεση σε βάρος της εβραϊκής κοινότητας πέρυσι στην ίδια πόλη είχαμε δεύτερη επίθεση σε βάρος ε, βουλευτού της Bundestag αφρικανικής καταγωγής και την προηγούμενη εβδομάδα στις εκλογές στη Θορυγγία γίναμε μάρτυρες ε, ε, του σπασίματος ενός ταμπού όταν υπήρξε συμμαχία με ένα λαϊκιστικό κόμμα για το σχηματισμό της κυβέρνησης. Την προηγούμενη εβδομάδα, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, υπήρξε μια παράσταση με ρατσιστικό περιεχόμενο ε, και δεν ε, λήφθησαν υπόψη ε, οι διαμαρτυρίες ε, ορισμένων ηθοποιών που δεν ήθελαν να γίνει αυτή η παράσταση. Δυστυχώ, ε, είμαστε ακόμη Αφρικανική Καταγωγή θύματα ρατσισμού, μυσαλλοδοξία, μίσου. Ε, κυρία συνάδελφε, παρακαλώ, έχετε, έχετε περάσει το χρόνο σας. Πρέπει να εφαρμόσουμε ε, τις αρχές της ισότιμης μεταχείρισης και θα πρέπει η αναξιοπρέπεια να τη βάλουμε σε πρώτη γραμμή. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λεμπρετό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο αντισημιτισμός αυξάνει στην Ευρώπη. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, η έκθεση 2019 του Υπουργείου Εσωτερικών αναφέρει αύξηση 74% των αντισημιτικών δράσεων. 34% των Εβραίων που ζουν στη Γαλλία νιώθουν ότι απειλούνται. Πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό το ανησυχητικό φαινόμενο. Αλλά για να αντιμετωπιστεί, πρέπει πρώτον να συνειδητοποιήσουμε ότι σήμερα υπάρχουν τρει πηγέ αντισημιτισμού. Πρώτον, υπάρχει ο αντισημιτισμό τη άκρα δεξιά, που είναι ο πιο παλιό, παραμένει. Στη συνέχεια υπάρχει κάτι πιο νέο, ο αντισημιτισμό τη άκρα αριστερά, που απορρέει από την αντισιωνιστική ιδεολογία. Και τρίτον υπάρχει ο Ισλαμιστικό ε, αντισημιτισμό που αυξάνεται στη Δυτική Ευρώπη εξαιτία τη αξέλεκτη μετανάστευση. Αυτό ακριβώ είναι που μου φαίνεται το πιο επικίνδυνο από τα τρία. Το αφήνουμε χωρί να αντιδρούμε. Σήμερα πρέπει να σταματήσει αυτή η ανοχή και να την αντιμετωπίσουμε χωρί να επιδείξουμε καμία δυναμία. Ε, τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Η αύξηση του αντισημιτισμού και η αύξηση του συναισθήματος ανασφάλειας όσον αφορά τους Ευρωπαίους Εβραίου είναι μεγάλη ήττα για τη σύγχρονη Ευρώπη. Οι Ευρωπαίοι πολιτικοί λένε ιστορίες για την προστασία των μειονοτήτων, αλλά οι περισσότεροι στις εβραϊκές κοινότητες σκέφτονται ότι πρέπει να φύγουν από την Ευρώπη, να μεταναστεύσουν. Αυτό είναι ένα πραγματικό παράδειγμα της ευρωπαϊκής υποκρισίας και δυστυχώ δεν είναι το μοναδικό. Κάποιες ομάδες των κοινωνιών μας έχουν γίνει πιο ίσες από άλλες. Και ενώ ε, θρυνούμε για τη μοίρα εκείνων που σε μεγάλο βαθμό εξαρτώνται από την υποστήριξη του κράτους, πιο επιτυχείς κοινότητες, όπως είναι οι εβραϊκές κοινότητες, αγνοούνται εντελώς. Η αύξηση του αντισημιτισμού επίσης είναι και μια ήττα της ευρωπαϊκής πολιτικής για την ένταξη και τη μετανάστευση. Άφησε να εισαχθεί εξτρεμισμό στην ευρωπαϊκή επικράτεια και θα πρέπει να θέσουμε τέρμα σε αυτό. Έχουμε χρόνο ακόμα έχουμε μεγάλη παράδοση. Εδώ πέρα έχουμε την ξενοφοβία με βία. Εμείς απορρίπτουμε τον ιστορικό ρεβιζιονισμό. Δεν επιτρέπουμε να χειραγωγείται ο αγώνας κατά του ασημιτισμού για να τα βάλουμε με αυτούς που τα βάζουν με τις παρανομίες που κάνει η Ισραηλινή κυβέρνηση σε βάρος των Παλαιστινίων. Δεν μπορούν να μας κατηγορούν αυτοί οι οποίοι είναι κατά των ε, πολιτικών ε, του Ισραήλ. Η ελευθερία και η δικαιοσύνη είναι πράγματα τα οποία υποστηρίζουμε και το κάνουμε αυτό καταδικάζοντας ακριβώς την κυβέρνηση του Ισραήλ αλλά και τον ε, κύριο Τραμπ και τι συμφωνίε τη διεθνή οι οποίες δεν σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μην μπερδεύουμε του θύτες με τα θύματα. Υπάρχει σιωνιστικό καθεστώς στο Ισραήλ και είναι αυτό που φταίει για τα όσα συμβαίνουν. Κύριος Μπότος, τελευταίος ε, και καλύτερος. Ευχαριστώ πολύ τι βρίσκεται στη βάση για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού και του μίσους. Πρέπει να το δούμε και σίγουρα χρειάζονται στρατηγικές και συγκεκριμένες πολιτικές. Οι πολιτικές αυτές όμως πρέπει γρήγορα να αναπτυχθούν και σε όλα τα κράτη-μέλη, στις πρωτεύουσες αλλά και στα χωριά χωρίς μια γενικευμένη εφαρμογή θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα που είχαμε στιωτητού στην ε, ε, ε, Ρουμανία όπου δύο μάγειρες ασιατικής καταγωγής χρειάστηκε να αλλάξουν δουλειά γιατί κάποιοι θεωρούσαν δεν μπορούσαν να τους βλέπουν τους ξένους αυτούς ανθρώπους εκεί. Οι δύο μάγειρες λοιπόν ουσιαστικά αναγκάστηκαν να ασχοληθούν με κάτι πολύ χαμηλότερο των δεξιοτήτων τους. Αυτό είναι απαράδεκτο, αλλά πλέον δεν είμαστε στο μεσαίωνα. Και πρέπει να αποφύγουμε να γυρίσουμε στις εφρικαλότητες του παρελθόντος. Ευχαριστώ, Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Επανερχόμεθα στην Αντιπρόεδρο, την κυρία Γιούροβα. Έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, σας είμαι ευγνώμων για την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το θέμα αυτό. Θα ήθελα να αντιδράσω σε διάφορα σχόλια που ακούστηκαν. Πράγματι, αναφερθήκατε στη βολιδοσκόπηση της Υπηρεσίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και του Ευρωβαρομέτρου, που πραγματικά τα στοιχεία δείχνουν ανησυχητικά και συγκλονιστικά στοιχεία. Όταν ρωτάτε έναν Εβραίο πολίτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ποια είναι η βασική του ή η βασική της ανησυχία, της είναι ασφάλεια. Όταν ρωτάς Ευρωπαίους που δεν είναι εβραϊκής καταγωγής, σας λένε ανησυχούμε για την υγεία μας, για τη δουλειά μας, για την οικογένειά μας. Και αυτό πράγματι είναι πολύ ανησυχητικό το ότι οι Εβραίοι έχουν τέτοιο θεμελιώδη φόβο να αντιμετωπίσουν. Και έτσι σχεδιάζουν να φύγουν από την Ευρώπη. Οι Εβραίοι που φεύγουν από την Ευρώπη ποτέ δεν ήταν καλό σημάδι. Και αυτή δεν είναι μια Ευρώπη που θέλουμε. Η κυρία Ρίς νομίζω που ήδη έφυγε ρώτησε κατά πόσο κάνουμε αρκετά. Με τα θλίψεις μου λέω όχι. Δεν κάνουμε ακόμα αρκετά και όλοι μας έχουμε υποχρέωση να κάνουμε πολλά περισσότερα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάστηκε σκληρά. Προσπαθούσα να επιτύχει απτά αποτελέσματα στην καταπολέμηση του αντισημιτισμού. Αποφασίσαμε να προωθήσουμε την οθέτηση του ορισμού για τον αντισημιτισμό που χρησιμοποιείται και από τα περισσότερα κράτη-μέλη. Ανοιχτά ομιλούμε και απευθυνόμεθα κατά των πηγών αντισημιτισμού αναφέρθηκε και εδώ, είναι η άκρα δεξιά, η άκρα αριστερά, οι Ισλαμιστές ριζοσπαστικοί ε, και διάφορες ε, συνωματικές θεωρίες. Γι' αυτό παροτρύναμε τα κράτη-μέλη, τους Υπουργούς Εσωτερικών, να εθετήσουν αποφάσεις για τη δημιουργία στατηγικής επίπεδο κατών μελών, στατηγικές κατά του αντισημιτισμού με συγκεκριμένα προγράμματα και σχέδια, κυρίως στον τομέα της ασφάλειας και στον τομέα της παιδείας. Οι στρατηγικές τώρα βρίσκονται στη διαδικασία δημιουργίας και επί γερμανικής προεδρίας θα εξετάσουμε τις στρατηγικές και θα αποφασίσουμε για την περαιτέρω πορεία. Θέλουμε να δούμε συγκεκριμένα μέτρα που θα συνοδεύονται από χρήματα για την ασφάλεια. Είναι απαράδεκτο πραγματικά οι εβραϊκές κοινότητες να χρηματοδοτούν την ασφάλειά τους και προστασία χώρων όπως είναι οι συναγωγές και τα σχολεία, να τα πληρώνουν οι Εβραίοι. Πρέπει να κάνουμε πολλά περισσότερα για την παιδεία. Και αυτό πρέπει να αντικαθοπτρίζεται και στι εθνικέ στρατηγικέ και πρέπει αυτά να συνοδεύονται τα προγράμματα από τα χρήματα. Και εδώ αναφέρονται και τα ευρωπαϊκά χρήματα. Έχουμε προβλέψει συγκεκριμένα ποσά για την παιδεία στον τομέα. Επίσης πήγα στο Auschwitz πριν από 15 μέρες την επέτειο των 75 ετών από την απελευθέρωση των ανθρώπων από το στατόπεδο και άκουγα τις αυθεντικές μαρτυρίες των επιζησάντων. Δεν θα μπορέσουμε να ακούμε μαρτυρίες από αυθεντικούς ανθρώπους πλέον πολύ σύντομα. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να εξηγούμε στις νέες γενιές τι ήταν το ολοκαύτωμα και να αλλάξουμε το αφήγημα, διότι Συνεχώς συζητούμε για τα αποτελέσματα του ολοκαυτώματος, τα φρικτά στατιστικά στοιχεία. Θα πρέπει όμως να αρχίσουμε σοβαρά να μιλάμε για τις πηγές, για τις ρίζες του ολοκαυτώματος. Που ξεκίνησε το ολοκαύτωμα. Γιατί ο Μάριαν Τούλς και αυτό ανέφερε στο Auschwitz-Birkenau στην τελετή. Δεν μίλησε για το παρελθόν, μίλησε για το παρόν. Πώς μπορεί να ξανασυμβεί Κάτι αθώο θα φαίνεται σιγά σιγά, θα κινείται με αργούς ρυθμούς και μετά από την παθητική μας τάση θα τροφοδοτείται και θα γιγαντώνεται και από την αδιαφορία μας. Μας προειδοποίησε να μην είμαστε αδιάφοροι. Τελευταίο σχόλιο όσον αφορά τις παρεμβάσεις σας για τις ομιλίες μίσου στο διαδίκτυο. Έχουμε μια συμφωνία με τους μεγάλους φορείς τη ψηφιακή να αφαιρούνται οι ομιλίε μίσου. Μπορεί αυτό να μην αρκεί. Θα πρέπει να έχουμε την αρχή εγκλήματο και τιμωρία και στο διαδίκτυο. Παρότρινα ένθερμα λοιπόν τι αρχέ επιβολή του νόμου σε όταν κράτη-μέλη να κυνηγήσουν τι διάφορε περιπτώσει, να αποδείξουν ότι δεν είναι δυνατόν να βασίζεται κανείς μόνο να, μην, να παραμένει εντύπωση δεν υπάρχει νόμο στο διαδίκτυο. Πρέπει να κάνουμε πολλά περισσότερα. Οι φορείς του νόμου έχουν δραστηριοποιηθεί περισσότερο. Αλλά μου λένε συνεχώς οι εκπρόσωποι των δυνάμεων τάξης ότι στην Ευρώπη του 21ου αιώνα το έγκλημα δεν έχει σύνορα, ο ψηφιακό χώρος δεν έχει σύνορα και οι αστυνομικέ αρχέ εμποδίζονται από τα εθνικά σύνορα και δεν μπορούν να κυνηγήσουν τα στοιχεία που θέλουν για τα διάφορα εγκλήματα και να πάνε στο άλλο κράτο μέλο. Και γι' αυτό θα ήθελα να σα ζητήσω να επανεξετάσετε τον κανονισμό για ηλεκτρονικά στοιχεία που ανέπτυξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διότι εάν υιοθετηθεί αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ στο να μπορέσει να διωχθεί το έγκλημα όπου αυτό διαπράτεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε, κύριε Αντιπρόεδρε. Και τώρα, εκ μέρους της Κροατικής Προεδρίας, το λόγο έχει η κυρία Νικολίνα Μπέρνιατς. Ευχαριστώ, ε, σας ευχαριστώ ε, για την συζήτηση. Σίγουρα και το Συμβούλιο Σύσσωμο είναι κατά οποιασδήποτε μορφή ρατσισμού, αντισημιτισμού και ρητορική μίσου. Έχουμε νομικό πλαίσιο, θα πρέπει να το εφαρμόσουμε και εμπράκτο. Αλλά θα πρέπει να εθετήσουμε και μέτρα για να προλάβουμε αυτή τη μυσαλλοδοξία. Χάρη στην παιδεία και σε καλή συνεργασία και αντίλογο στη συζήτηση. Το Συμβούλιο θα παρακολουθεί εκ του αυτά τα θέματα, λαμβάνοντα υπόψη όλα τα σχόλια των Ευρωβουλευτών, όπω προέκυψαν στη σημερινή συζήτηση. Σα ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ τους συναδέλφους ε, για τη συμμετοχή τους ε, και τον ε, καλό τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης και να ολοκληρώσουμε αυτό το θέμα, έχω και μία ανακοίνωση πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα. Η ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ανακοίνωσε στον πρόεδρο τις αποφάσεις για την τροποποίηση της σύνθεσης των επιτροπών, απόφαση που θα δημοσιευθεί στα σημερινά πρακτικά και θα τεθεί σε ισχύ από τη μέρα της ανακοίνωσης. Και περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης που προβλέπει δήλωση του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την συνεχή απειλή κατά του κράτους δικαίου στην Πολωνία. Να σας ενημερώσω ότι για τις μπλε κάρτες και το Catch the Eye γνωρίζετε τη διαδικασία, οπότε δεν χρειάζεται άλλες εξηγήσει. Να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο του Συμβουλίου και της Κρατικής Προεδρίας, την κυρία Μπέρνιατς. Τα μέλη θα ήθελα να τονίσω για άλλη μια φορά ότι το κράτος δικαίου παίζει ε, σημαντικό ρόλο σε όλα τα κράτη-μέλη. Το κράτος δικαίου αποτελεί εγγύηση ότι τηρούμε τα τις βασικές μας αξίες. Θεωρώ ότι το κράτος ε, δικαίου δεν μπορούμε να το δούμε ανεξάρτητα. Πρόκειται για έναν κρίκο ενός γενικότερου συστήματος. Είναι κοινή ευθύνη των θεσμικών οργάνων και των κρατών ε, μελών να ενισχύσουν το κράτος δικαίου, το οποίο να αποτελέσει τον θεμελιώδη λίθο του συστήματός μας. Επίσης αυτό σημαίνει ανεξαρτησία των δικαστικών αρχών έτσι ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει πολύ καλά το κράτος δικαίου και να υπάρχει και ασφάλεια δικαίου. Δυνάμει του άρθρου 7 έγιναν τρεις ακροάσεις τον Ιούνιο, Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο του 2019 στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων για να δούμε τις εξελίξεις στην Πολωνία. Επίσης έχει γίνει ενημέρωση για την εξέλιξη της κατάστασης το 2019 τον Φεβρουάριο, Απρίλιο, Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο. Τώρα η Προεδρία θα συνεχίσει την διαδικασία στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων. Επίσης γίνεται διάλογος σε πολιτικό επίπεδο για να δούμε ποια είναι τα απτά αποτελέσματα ως προς την εξέλιξη της κατάστασης στην Πολωνία. Ευχαριστούμε την αντιπρο... και τώρα η Αντιπρόεδρος κυρία Γιούροβα. Προέδρε, αξιότιμα μέλη. Θα θυμάστε ότι στις 15 Ιανουαρίου ε, ο Επιτρόπος Ρέντερς και εγώ σας ενημερώσαμε για την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Πολωνία. Έκτοτε είμαστε σε επαφές με τις πολωνικές αρχές. Ο Επίτροπο Ρέντερς επίσης ε, συνάντησε στις 24 Ιανουαρίου τους εκπροσώπους της δικαιοσύνης. Το ίδιο έκανα και εγώ στις 25 Ιανουαρίου. Με την ευκαιρία αυτή ε, συναντήθηκα με τους ε, Προέδρου του Ισάνο και Κάτω Βουλής, ε, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον Πρόεδρο του Συνταγματικού Δικαστηρίου και τον, Ευρω... τον Συνήγορο του Πολίτη. Άκουσα προσεκτικά τα επιχειρήματα της πολωνικής κυβέρνησης και τους εξήγησα τη στάση της Κομισιόν. Η Κομισιόν είναι έτοιμη και διαθέσιμη να επιλύσει το ζήτημα με κάθε διαθέσιμο τρόπο. Επίσης, πάντοτε θα, εκπληρώσει, θα εκπληρώνει το ρόλο της ως θεματοφύλακας των συνθήκων. Έτσι λοιπόν δεν θα διστάσει να χρησιμοποιήσει τις διαδικασίες επί παραβάση όποτε υπάρχουν ζητήματα συμβατότητας στην Ένωση. Αντιστοίχως το, η διαδικασία του άρθρου 7 συνεχίζει ε, διότι η κατάσταση θέτει συστημικό, συστημική απειλή εναντί του κράτους δικαίου. Επίσης ε, υπάρχει ε, αυτή τη στιγμή το νομοσχέδιο ε, το οποίο αφορά στην ε, λειτουργία του δικαστικού σώματος. Εξήγησα ότι η ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος είναι αυτό που κάνει την Κομισιόν να ανησυχεί. Γι' αυτό το λόγο έστειλα στις 19 Δεκεμβρίου 2019 ένα σημείωμα, μια, μια επιστολή στις πολωνικές αρχές ε, ζητώντας να ενισχυθεί το κράτος δικαίου προλαμβάνοντας τα προβλήματα και εργαζόμενοι ως προς την πύλησή τους κάθε φορά που αυτά προκύπτουν. Επίσης κάλεσα όλα τα κρατικά όργανα να μην προχωρήσουν τις διαδικασίες ε, για το νέο νομοσχέδιο πριν γίνουν οι απαραίτητες διαβουλεύσεις. Στις 16 Ιανουαρίου η Κομισιόν επίσης ε, εξέδωσε ε, μία σύσταση ε, αναφέροντας τις ανησυχίες της. Στις 24 ε, Ιανουαρίου εγκρίθηκε η νέα νομοθεσία και στις 4 Φεβρουαρίου κυρώθηκε ο νόμος από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αυτός ο νόμος μας δίνει μια σειρά θεμάτων που μας κάνουν να ανησυχούμε. Για παράδειγμα, μπορεί περαιτέρω να υποσκάψει την ανεξαρτησία των δικαστών στην Πολωνία. Μας κάνει να ανησυχούμε για τη συμβατότητά του με την ευρωπαϊκή νομοθεσία επιπλέον. Και εμείς εξετάζουμε αυτά τα ζητήματα λεπτομερώς. Σας διαβεβαιώ ότι είμαστε ε, έτοιμοι να πάρουμε κάθε μέτρο που θα διασφαλίσει ότι θα έχουμε συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Επίσης, στις 15 Ιανουαρίου, το Ανώτατο Δικαστήριο έβγαλε δύο αποφάσεις, ε, εφαρμόζοντας ε, μια προκαταρκτική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σχετικά με την ανεξαρτησία του πειθαργικού. Και ε, στις 5 Δεκεμβρίου επικυρώθηκε αυτή η απόφαση δηλώνοντας ε, πως το πειθαρχικό σώμα δεν είναι ένα ανεξάρτητο σώμα ε, εντός, ε, μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και της Εθνικής Νομοθεσίας. Επίσης, στις 23 Ιανουαρίου το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε ότι οι δικαστές που είχαν διοριστεί από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο δεν πρέπει να αποφασίζουν. Επίσης, όλες οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου ε, επικυρώθηκαν. Μια άλλη εξέλιξη είναι ότι το συνταγματικό δικαστήριο έχει λάβει μία προσφυγή σχετικά με την ανεξαρτησία των δικαστών. Ε, αυτό μετά από την προκαταρκτική απόφαση στις 19 Νοεμβρίου του 2019. Στις 28 Ιανουαρίου του 2020 το Συνταγματικό Δικαστήριο πήγε, πήρε μία απόφαση που είχε ε, στόχο να ανασταλεί η εφαρμογή της απόφασης ε, του πειθαρχικού. Επίσης, στις 24 Ιανουαρίου, αν θυμάστε, είχε ζητήσει η Επιτροπή να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα έτσι ώστε να σταματήσει η λειτουργία του πειθαρχικού. Στο μεταξύ, παρατηρώ απλώς ότι το Πειθαρχικό Συμβούλιο ε, συνεχίζει να λειτουργεί. Με λύπη μου λοιπόν παρατηρώ αυτές τις πρόσφατες εξελίξεις ε, οι οποίες είναι ιδιαίτερα σοβαρές. Αυτό αντικατοπρίζεται και στην πρόσφατη ε, απόφαση της κοινοβουλευτικής ε, συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης που μιλά για την λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών και το κράτος δικαίου στην Πολωνία. Ταυτόχρονα Ήθελα να επαναλάβω ότι η Επιτροπή παραμένει έτοιμη να συνεχίσει τον διάλογο με τις πολωνικές αρχές ώστε να επιληθούν τα ε, ζητήματα που είναι ανοιχτά. Επίσης, ε, ε, θέλουμε ο διάλογος